Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, μία ακόμα ε, ταπεινωτική ε, έκκληση για το άρθρο 50. Έχω μια λύση. Άκουσα κύριε Μπαρνιέ, που είπατε προηγουμένω ότι αν αυτή η συμφωνία αποχώρηση ε, περάσει, το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων μπορεί να διαρκέσει έω και τέσσερα χρόνια. Όχι, φτάνει. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε άλλα τέσσερα χρόνια ε, τη ζωή μα, τέσσερα χρόνια αγωνία. Ούτε εσεί θέλετε να σπαταλήσετε αυτά τα χρόνια. Έχετε ένα σχέδιο. Θέλετε τι Ηνωμένε Πολιτείε Ευρώπη. Θέλετε το στρατό σα να μπουν όλοι στην Ευρωζώνη. Να καταργηθούν τα κράτη-έθνη. Εμεί είμαστε απλώ ε, κάτι το ενοχλητικό. Και όπω είπε ο κ. Βερχόφσταντ για τι ευρωεκλογέ, δεν θέλετε να έρθω εγώ και όλοι οι άλλοι ευρωσκεπτικιστέ να ξαναγυρίσουν στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια πολύ απλή λύση λοιπόν το Βρετανικό αίτημα παράτασης ε, να έρθει αντιμέτωπο με βέτο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να φύγουμε στις 29 Μαρτίου. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες προετοιμασίες έχουν ήδη γίνει. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες αναταράξεις μέχρι τότε, θα φύγουμε και εσείς και εμείς θα συνεχίσουμε τις ζωές μας. Μόνο αυτή η καλή λύση υπάρχει μπροστά μας. Από το ENF. Ο κύριος Μπάτεν. Η κυρία Μέη μπορεί να είναι εντελώς ανίκανη, αλλά ακολουθεί ένα σχέδιο από την αρχή. Το σχέδιο ήταν να καθυστερήσει τον Brexit, να τον παρεμποδίσει και τέλος να τον ατρέψει. Όλη η διαδικασία της αποχώρησης βασίστηκε σε ψεύτικα επιχειρήματα. Το βασικό ήταν ότι δεν μπορούμε να φύγουμε χωρίς μια, τιμηθική καλή συμφωνία. Η συμφωνία είναι άθλια και την έχει απορρίψει η Βουλή των Κοινοτήτων. Όχι γιατί ήταν κακή, αλλά γιατί δεν ήταν αρκετά κακή για αυτού. Αργότερα, σήμερα, το Κοινοβούλιο θα απορρίψει και την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, το no deal. Και την Πέμπτη θα ψηφίσει μάλλον υπέρ μια παράτασης του άρθρου 50. Αλλά γιατί. Ο κύριος Γιούγκερ είπε στην κυβέρνησή μας, σαν να είμαστε σχολιαρούδια, ότι δεν θα υπάρξει τρίτη ευκαιρία για διαπραγμάτευση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κοινοβούλιο που δεν θέλουν να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σκοπεύει να προδώσει τη δημοκρατική απόφαση του δημοψηφίσματος. Ο κύριος Τίμερμανς εξέφρασε την αγανάκτησή του γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε την ε, συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Τίμερμαν είπε ότι μόνο το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να δώσει κατεύθυνση, καθοδήγηση σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν είναι σωστό. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν μπορούν να καθοδηγήσουν τη διαδικασία. Όταν η Βουλή των Κοινοτήτων ζητήσει παράταση του άρθρου 50, τότε πρέπει να την απορρίψετε. Το άρθρο 50 λέει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 29 Μαρτίου, τότε οι συμφωνίε αυτόματα πάβουν να ισχύουν μην κάνετε τίποτα. Και θα εξασφαλίσετε ότι θα πεταχτεί έξω στις 29 Μαρτίου το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το καλό σας, για το καλό μας, διώξτε μας με σκλωτσιές. Πρέπει να είμαι πιο αυστηρή με τον χρόνο ομιλίας, διότι ξεπερνάμε το χρόνο μας. Κύριε Ντότζ, ε, κύριε είμαι βέβαιη ότι θα περιοριστείτε στο ένα λεπτό σας. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χθε το βράδυ, οι βουλευτέ όλων των κομμάτων ε, καταψήφισαν ε, την συμφωνία. Λυπάμαι που δεν έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδο στο θέμα αυτό. Η συμβουλή του Ανώτατου Νομικού Συμβούλου είναι σαφής. Ο νομικός κίνδυνος παραμένει χωρίς να αποδεικτικά στοιχεία της κακής πίστης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχει δυνατότητα να ξεφύγει από τον μηχανισμό ασφαλείας, τον backstop. Η θέση μας είναι σαφής. Θέλουμε συντεταγμένη αποχώρηση, θέλουμε μία λύση που να λειτουργεί καλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τους πιο κοντινούς γειτόνους μας, τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Μια τέτοια συμφωνία όμως θα πρέπει να σέβεται την ε, συνταγματική ακαιρεότητα της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω σε κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν. Αναφέρθηκαν επανειλημμένα τα δικαιώματα των πολιτών. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει αυτό να είναι διαπραγματευτικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις. Η Βουλή των Κοινοτήτων ήδη είπε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών σε κάθε ενδεχόμενο. Ε, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι και όχι να μιλάμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ κύριο Λεβαντόφσκι, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπώ την γεωργική παραγωγή της Βρετανίας, αλλά το Brexit δεν μ' αρέσει. Με κατάπληξη ε, συγκλονισμένος παρακολουθώ αυτά που συμβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παλαιότερα λέγαμε ότι ε, τα πρώην κομμουνιστικά μέρη της Ευρώπης ε, ψάχνουν για κάποιο πρότυπο, αναζητούν κάποιο πρότυπο και ένα τέτοιο πρότυπο ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσο ε, μεγάλος ήταν τότε ο θαυμασμός μας, τόσο μεγάλη είναι σήμερα η απογοήτευσή μας. Βλέπουμε να παίζονται πολιτικά παιχνίδια χωρίς να γίνονται προσπάθειες για μια επικοδομητική λύση. παίζονται διάφορα πολιτικά σενάρια, καταψηφίζονται οι προτάσεις που βρίσκονται επί τάπητο. Πρέπει όμως να σκεφτούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ε, όλα αυτά σημαίνουν αβεβαιότητα για πολλού πολίτες και ακόμα για πολλούς Πολωνούς που αναζήτησαν καλύτερη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν γνωρίζουμε πώ θα μπορέσει να βρεθεί λύση τώρα, εφόσον δεν βρέθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Στο, στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και κατά τη παραπληροφόρησης. Το Βρετανικό δημοψήφισμα τροφοδοτήθηκε από πολλές ε, ε, λανθασμένες ψευδείς πληροφορίες από ε, την Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν ε, το επικίνδυνο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα της κυβερνοασφάλειας και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Γουαλτιέρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για δεύτερη φορά η Βρετανική κυβέρνηση δεν κατάφερε να διασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ήταν μεγάλο σφάλμα που δεν προσπάθησαν ε, να συνενώσουν όλες τις ε, πολιτικές ε, δυνάμεις προς το συμφέρον της χώρας. Αντιθέτως, η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να πάει με το μέρος των υπέρμαχων της αποχώρησης. Κάτι το οποίο γύρισε μπούμερανγκ και το είδαμε αυτό χθες. Κύριε Χένκελ, λάθος κάνατε. Όπως είπε ο κύριος Μπαχνιέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν Δίκαιο, διαφανής και επικοδομητικός εταίρος αυτή τη διαπραγμάτευση. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε τη συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με προστασία των πολιτών. Να σας πω τώρα ότι έχουμε ξεκάθαρο ε, καθήκον να προστατεύσουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σε αυτή τη διαδικασία και να ε, διασφαλίσουμε διατηρήσουμε και την ενευτική διαδικασία στην ε, Ιρλανδία. Λαμβάνοντα υπόψη βέβαια και τι ε, κόκκινε γραμμέ τη Βρετανική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η μοναδική συμφωνία αποχώρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή και μόνο αυτή μπορεί ε, να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι γίνεται από εδώ και πέρα ελπίζουμε να απορριφθεί η πρόταση του No Deal που θα ήταν καταστροφική για τον Βασίλειο. Δεύτερον, χρειαζόμαστε σαφεί κατευθύνσει για το πώ να αποφύγουμε με αυτά βήματα το σενάριο του No Deal. Όσο πιο. Ε, μια, πιο στενή συνεργασία βάσει τη τελωνική συνεργασία θα είναι επωφελή και για τι οικονομίε μα, αλλά θα διασκεδάσει και τι ανησυχίε για τον backstop. Πρέπει να αφήσουμε τα μικροπολιτικά και να εργαστούμε επικοδομητικά προς όφελος ε, των ε, πολιτών. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό και εφικτό, η μοναδική εναλλακτική θα είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στο λαό να αλλάξει η κυβέρνηση ή να πει όχι στο Brexit. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να κάνουμε. Όχι μια συζήτηση για τη διάρκεια τη παράταση. Γιατί για εμά είναι σαφέ ότι η παράταση είναι ένα εργαλείο. Και όλε οι επιλογέ τίθενται επιτάπητο, αρκεί να υπάρχει ε, εύλογη τεκμηρίωσή του με σαφή προοπτική. Και εμεί θα είμαστε ανοιχτοί και υπεύθυνοι και απέναντι στους Βρετανούς πολίτες που παραμένουν Ευρωπαίοι πολίτες. Συνάδελφοι, είναι δύσκολη συζήτηση, το ξέρω. Και οι συνάδελφοι θέλουν να εκφράσουν τα επιχειρηματά τους σαφώς, αλλά είμαι υποχρεωμένη να σας πιέσω γιατί έχουμε και πολλές ψηφοφορίες. Ε, κύριε Νίκολσον, 1,5 λεπτό ακριβώς, μην με απογοητεύσετε. Άκουσα σήμερα το πρωί, με βαριά καρδιά, όλα όσα υπόθηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο. Και τίποτα θετικό δεν άκουσα να λέγεται. Όλα αρνητικά ήταν. Όλοι είναι στα χαρακόμματα, τίποτα επικοδημητικό δεν βγαίνει το στόμα τους. Ο κύριος Τίμερμανς είπε, εδώ φτάσαμε, οι λύσεις πρέπει να έρθουν από το Λονδίνο. Κύριε Τίμερμανς, εσείς και ο κύριος Γιούνκερ δεν παίξατε κάποιο ρόλο και δεν πρέπει επομένω, εφόσον παίξετε ρόλο, να, βρείτε, να είσαστε και θύμα τη λύση. Επίση, κάποιοι, κυρία Ζήμερ, ε, έβγαλε τη γάτα από το σάκο για τη Βόρεια Ιρλανδία. Υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν θέλουν, ακόμα και αυτά που δεν θέλουν το δημοψήφισμα για, το, για τα σύνορα, δέχονται τη συμφωνία της α, ε, Μεγάλης Παρασκευής. Κύριε Μπαρνιέ, είπατε ότι η μόνη ευθύνη βαραίνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αμπά και εσάς και εσεί έχετε τρομερές ευθύνε. Δεν αρκεί να έρχεστε σε επαφή μόνο με Βορειοϊρλανδού που σας λένε αυτά που θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν και άλλες φωνές στη Βορειοϊρλανδία. Και θα πρέπει να ακούσετε και τις άλλες φωνές. Ζητώ συγγνώμη που σας τα λέω αυτά. Με κάθε σεβασμό σας τα λέω. Αλλά είναι γεμάτη ελαττώματα η συνθήκη σας και δεν πρέπει να λειτουργήσει. Χρειαζόμαστε κάποιο άλλο τρόπο. Χρειαζόμαστε παράταση ε, του άρθρου 50 για να βρούμε αυτόν τον άλλο τρόπο. Και δεν αρκεί να μας λέτε ότι πρέπει να έχουμε αιτιολόγηση για την παράταση. Θέλουμε παράταση για να βρούμε μια καλή συμφωνία. Γιατί ο λαό μου και οι άνθρωποι που εκπροσωπώ θέλουν καλή συμφωνία. Κύριε Μπαγνιέ, σήμερα το πρωί είπε ότι όλα τα αγαθά, υπόθηκε ότι όλα τα αγαθά που πηγαίνουν από την ε, Ιρλανδία στη Βόρεια Ιρλανδία θα περνάνε απρόσκοπτα. Το είπαν αυτό σήμερα το πρωί στην Ιρλανδία. Μπορείτε να το πείτε εσείς αυτό εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Φοβάμαι όμως ότι αποτύχατε όσον αφορά την τήρηση του χρόνου. Η κυρία Χάρκιν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Πρωθυπουργό, η κυρία Μέη, ε, είναι δυσαρεστημένη με την ήττα της, αλλά εγώ όπως και πολλοί από εσά λυπούμε που φαίνεται ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχει χάσει το δρόμο του. Ε, είδαμε πολλές διαφορετικές απόψεις κατά τη διάρκεια των ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι αυτό που έχει σημασία είναι το μέλλον και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το 1992 η Δανία, το 2001, το 2008 η Ιρλανδία, το 2005 η Γαλλία και οι κάτω χώρες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είπανε όχι σε διάφορες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Ναι, ως ε, μεμονωμένες χώρες και ως Ένωση, ε, ακούγοντας, ε, αφουγκραζόμενοι ε, και με διάλογο, οι πολίτες μας κατάφεραν να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσουν. Και παρά αυτόν που είπε ο κύριος Φαράς, πιστεύω ότι αυτό μπορεί ακόμα να γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Διαφωνώ βαθύτατα μαζί του όταν μιλάει για ε, οργή περιφρόνηση και ε, ακαμψία. Προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη για μια διαιρεμένη χώρα ε, στους ώμους άλλων. Συμφωνώ με τον Μισελ Μπαρνιέ ήμασταν και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε υπομονετικοί, ε, να υποστηρίζουμε και να έχουμε σεβασμό και ευχαριστώ την ομάδα του για την ε, δουλειά που έχει κάνει. Και τέλος, ε, στον κύριο Γκουαλτιέρη να πω ότι η παράταση είναι ένας τρόπος να βρούμε έναν τρόπο και πρέπει να εξερευνήσουμε ακόμα όλες τις επιλογές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Εύαν, σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε γίναμε μάρτυρες ακόμα μιας ε, τεράστιας ήττας για την Βρετανική κυβέρνηση σε μια ψηφοφορία που θα ήταν, για μια συμφωνία που θα ήταν καταστροφική για την Ουαλία. Θα την έβγαζε από την Ενιαία Αγορά και από την Τελωνιακή Ένωση. Είναι σαφές ότι το Βρετανικό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να καταλήξει κάπου. Γι' αυτό πρέπει να επιστρέψουμε στο λαό. Η συγκέντρωση πλούτου στο Λονδίνο ε, είναι αυτή που είναι υπεύθυνη ε, για όλο αυτό το χάλι. Και το Βρετανικό Κοινοβούλιο είναι αυτό που μα ε, κρατάει μέσα σε αυτό το χάλι. Η δημοκρατία είναι η λύση. Πρέπει να δώσουμε στο λαό ε, τη δυνατότητα να εκφραστεί για τελευταία φορά για το μέλλον του. Τώρα που έχουμε δει την πραγματική κατάσταση. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και όταν αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και οι απόψει του λαού. Αυτό είναι δικαίωμά του. Η Ουαλία αυτό ακριβώς έχει δείξει. Το 55% τώρα στηρίζουν το Remain μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2016. Χρειαζόμαστε παράταση του άρθρου 50 ε, και χρειαζόμαστε νέα ε, ψήφο για το λαό. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, η κυρία Άντερσον. Ο λαός της νήσου της ε, Ιρλανδίας έχει κουραστεί από την ανοργανωσιά και την αταξία. Η σαφής μας θέληση είναι να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αγνοηθεί. Το απόλυτο χάο του όχι μόνο χθε το βράδυ, αλλά καθ' όλη τη διαδικασία του Brexit, άφησε κοινότητε ή απόχνωση. Αυτή σε απόγνωση. Αυτή η φάρσα έχει σχεδιαστεί από του συντηρητικού και έχει παραδοθεί στους ε, Βόρειους Ιρλανδούς μέσω της διαίρεσης από τον DUP. Θεωρούμε ότι η συμφωνία αποχώρησης και το backstop που τη συνοδεύει είναι η λιγότερο κακή επιλογή που μπορούμε να δεχτούμε. Και αυτό έχει απορριφθεί πλήρως, ξανά από το βρετανικό πολιτικό κατεστημένο που κάνει ό,τι να είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη Συμφωνία τη ε, Μεγάλη Παρασκευή σε όλα τα τμήματά τη. Αυτό συμπεριλαμβάνει και, την, και το θεμητό, τη θεμητή δημοκρατική πορεία ε, προς την ε, Ιρλανδική ενοποίηση. Ο, η Βρετανίδα Πρωθυπουργό η ίδια πιστεύει ότι το Brexit αυξάνει την υποστήριξη για την ενοποίηση της Ιρλανδίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε τον Απρίλιο του 2017 ότι αν επανενωθεί η Ιρλανδία, τότε όλη η νήσος αυτόματα θα παραμείνει τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι πρέπει να ε, ετοιμαστούμε για ένα no deal για ένα κρασάρισμα. Ποιο μεσόαστα φρένα θα κάτσει σε ένα τρένο που πάει να πέσει στον κρεμό ή επίτηδε να εκτοχιαστεί. Επομένω, ο κόσμο θέλει να βγει από αυτό το τρένο, να κατέβει. Θέλουμε την Ένωση τη Ιρλανδία και κάνω έκκληση να υποστηρίξετε την διεξαγωγή ενό δημοψηφίσματο για την ενοποίηση τη ε, Ιρλανδία. Είναι δημοκρατικό κάτι τέτοιο. Βασίζεται στη συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή που θέλετε να τη στηρίξετε σε όλα τα τμήματά της. Η πρόεδρο διακόπτη θα πρέπει να ολοκληρώσετε το επιχείρημά σας μέσα στο χρόνο που έχετε. Ο κύριο Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η στιγμή να μιλήσουμε και να διαρωτηθούμε ποιοι είναι οι βαθύτεροι λόγοι του Brexit. Ακόμα και σήμερα ακούσαμε και εδώ τις δηλώσεις του Μακρόν όμως και του Γιούνκερ ε, όλου του κατεστημένου για τις ευθύνες ε, του Brexit. Ε, ότι υπάρχουν πληροφορίε που μπέρτεψε τον ε, Βρετανικό λαό. Ο Βρετανικός λαός όμως ε, με τα λόγου γνώσεως αποφάσισε να μην πει στο ενιαίο νόμισμα. Αποφάσισε να μην δεχτεί το Σέγγεν, να μην δεχτεί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Πάντα αντέδρασε με τα λόγου γνώσεων κατά των πολιτικών της λιτότητας, κατά της Γάλλο-Γερμανικής Συμμαχίας. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Πρέπει να ε, σκεφτούμε και την ε, ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, απεικιοκρατική στάση Γαλλίας-Γερμανίας και τις πολιτικές λιτότητας. γιατί φοβάμαι ότι το Brexit θα είναι απλώς ένα επεισόδιο στη σειρά της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, κύριε Ατκίσον, ένα λεπτό. Ζητώ συγγνώμη για τα ψέματα που λένε οι πολιτικοί μας. Ο κύριος Σταγιάννη, ένας σταλός, λέει σε μια γερμανική εφημερίδα ότι ο Βρετανικός λαός δεν ήθελε τον Brexit. Στις εκλογές του 2017, η τεράστια πλειοψηφία των ε, Βρετανών ψήφισαν ε, υπέρ της αποχώρησης. Τώρα η κυρία Μέη καταψηφίστηκε η πρώτη της πρόταση, τώρα ε, ζητάει ψήφο για, μια, για ένα no deal. Ουσιαστικά σήμερα ε, μια συντηρητική θα ε, καταψηφίσει και θα κυρώσει το Brexit. Αλλά λένε οι εργατικοί ότι λένε ψέματα. Υπάρχει ένα άλλο κύκλο τη κολάσεω ε, όπου θα πάνε όλοι αυτοί. 29 Μαρτίου, λοιπόν, στην πλατεία μπροστά στο Κοινοβούλιο, ελάτε μαζί μου για να ξαναπάρουμε πάλι τον έλεγχο. Ο κύριο Βόλφ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Πριν δύο μέρες ε, διαγνώστηκε ε, μοιραία ασθένεια στον θείο μου και θα πεθάνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ε, πέρασε τη ζωή του προστατεύοντας ε, παιδιά από την κακοποίηση παιδόφιλους και το 2014 τον Ιούνιο ψήφισε να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πεθάνει χωρίς να δει το Brexit όμως λόγω μιας πολιτικής τάξης που περιφρονεί αυτόν και όλους τους ψηφοφόρους του ε, ε, της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν θέλουν να ακούσουν τους ψηφοφόρους που ήθελαν να παραγούν από αυτούς. Θα πεθάνει επειδή δεν θα δει το Brexit λόγω πολιτικών όπως είναι ο Τόνι Μπλερ που προσπάθησαν να σταματήσουν δημοκρατική ψήφο των ε, των Βρετανών. Ο θείο μου ελπίζω να ε, πεθάνει εν ειρήνη, αλλά για όλους τους ε, για όλους όσους επιβιώσουν να γνωρίζετε ότι ο Θεός δεν φαίνεται να είναι με το μέρος σας. Ο, Μπροκ, ο κύριος Μπροκ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μπούλμαν, κύριε Τίμερμανς, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχει νομίζω μια συμμαχία στην ένα συνασπισμό στην Βουλή των Κοινοτήτων που δεν ε, μπορεί ε, να παρουσιάσει κάποιο αποτέλεσμα. Ε, έχουμε αυτούς που θέλουν να παραμείνουν διότι ελπίζουν σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα και γι' αυτό είναι άκαμπτοι. Μετά έχουμε του φαράζ αυτού του κόσμου και έχουμε τους άλλους που ενεργούν με κομματικά κριτήρια. Ε, τρεις εργατικοί ε, υπερψήφισαν την συμφωνία και γι' αυτό δεν μπορεί η Βουλή των Κοινοτήτων ε, να βρει μια λύση. Τα δύο μεγάλα κόμματα θα πρέπει επιτέλους να συνομιλήσουν μεταξύ τους και θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχει κάποια πλειοψηφία που, με μια πρόταση που αξίζει να συζητήσουμε επικοδομητικά. Δεν θέλουμε να δώσουμε καμία παράταση χωρίς ε, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ε, το απλά να έχουμε μια παράταση μήπως και συμβεί κάτι δεν μου φαίνεται σωστό. Θα πρέπει η Βουλή των Κοινοτήτων λοιπόν να μας κάνει κάποια δήλωση, ε, να μας παρουσιάσει μια βάση με την οποία να μπορούμε να προχωρήσουμε. Τα τελευταία δύο-δυόμιση χρόνια διαπραγματευτήκαμε, αλλά χωρί κανένα αποτέλεσμα. Μισελ, σε ευχαριστώ θερμά για τη δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστώ ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που έχει κάνει. Ε, πιστεύω όμως ότι ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, ακροβατικά και πάλι δεν θα είχαμε πετύχει κάτι στο στη Βουλή των Κοινοτήτων, διότι υπήρχε αυτή η αρνητική στάση. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παρουσιάσει αποτελέσματα ούτω ή άλλω. Και όσον αφορά τα σύνορα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να μπει από την πίσω πόρτα στην ενιαία αγορά χωρίς να πληρεί τα κριτήρια της ενιαίας αγοράς. Οι δηλώσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί είναι κακόβουλες, λαϊκιστικές και δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Δηλαδή, ε, το να μπει ε, στα κρυφά ε, στην ενιαία αγορά είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ένα μισή λεπτό, κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Μπαγνιέ, κύριε Υπουργέ, λίγες μέρε πριν από την Σύνοδο Κορυφή υπάρχουν πολλά ερωτήματα και υπάρχουν δύο τουλάχιστον κρίσιμα για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit, καταρχά, και η ήττα χθε για την Μέη και η πιθανή παράταση του άρθρου 50 που είναι μάλλον απόφευκτη από ό,τι φαίνεται δεν θα πρέπει να μας κάνει να παρατείνουμε την αγωνία η οποία έχει ήδη χρονίσει από το 2016 μέχρι σήμερα. Οι συνάδελφοι από τη Βουλή των Κοινοτήτων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα βασικά θέματα, θα πρέπει να ξαναδώσουν το λόγο στους Βρετανούς πολίτες, να ακούσουν τη φωνή τους για να δουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε. Γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν ε, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο μόνος τρόπος είναι να ξαναδώσουν το λόγο στους πολίτες και να ακούσουν τη φωνή τους. Παρότι πολλοί από αυτούς φοβούνται, πολλοί από τους συνάδελφους μας που είναι υπέρ του Brexit ε, φοβούνται να δώσουν το λόγο στους πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα ακόμα πιο σημαντικό για το μέλλον της Ένωσης είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Θα υιοθετήσουμε μέτρα πολύ σημαντικά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε να τροποποιούμε τους κανόνες με τους οποίους λειτουργούμε. Θα πρέπει να παρέμβουμε στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει να βασίζεται σε οικολογικούς στόχους και στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να είναι ένα εξάμεινο λιτότητας, αλλά θα πρέπει να βασιστούμε στους στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Ο κ. Βαντάλεν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλημέρα. Η New Financial χθε ανακοίνωσε ότι πάνω από 250 επιχειρήσει ε, στον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν αποχωρήσει ή θα φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε λοιπόν μία ε, απώλεια 5.000 θέσεων και ένα δι ε, θα φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτία αυτών των κινήσεων. Αυτά είναι τα νούμερα που ξέρουμε, έτσι. Πέραν τούτου, δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι συνέπειε. Μια μεγάλη λοιπόν αλλαγή για το Μηνοβασίλειο, αλλά και από αυτή την πλευρά τη μάχη θα υπάρξουν σημαντικά πλήγματα από το Brexit ε, στην αλληλεία ή στι μεταφορέ, για παράδειγμα. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι στο Βρετανικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει καμία πλειοψηφία για καμία πτυχή του Brexit και αυτό κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε μια νέα προσέγγιση. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ένα new deal, όχι no deal. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, να, να κάνουμε μάλλον μια πρόταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία θα είναι αναγκασμένο να αποδεχθεί. Ευχαριστώ κύριε Φλάνναγκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ακούω τον όρο αλληλεγγύη να χρησιμοποιείται ξανά και ξανά. Η αλληλεγγύη βέβαια έχει πολλές μορφές ε, και από πολιτικής και από οικονομικής άποψης. Ο Επίτροπος ε, Τίμερμανς μίλησε για τη συνεχιζόμενη προετοιμασία για μια νέα συμφωνία. Ε, για τη δουλειά που έχει γίνει στην πράξη μέχρι τώρα. Αλλά ποιο είναι ο σχεδιασμό για την οικονομική στήριξη προ την Ιρλανδική οικονομία σε περίπτωση μη συμφωνία. Θα ήθελα μια πραγματική απάντηση. Η ελληνική μέχρι τώρα δεν ε, έχει μεταφραστεί σε κονδύλια στην ουσία. Όταν ε, μιλάμε για αλληλεγγύη, παράλληλα βλέπουμε ότι στην Ιρλανδία δανειστήκαμε και κάψαμε 3,5 δις ε, ε, πέρυσι κατόπιν εντολών της ΕΚΤ και πρέπει να τεθεί ένα τέλο σε αυτή την παράνοια. Κύριε, ε, κύριε Μπαρνιέ, είπατε ότι ε, παραμένετε ήρεμοι και με σεβασμό προ ε, τον λαό. Πράγματι, γιατί όσοι βρίσκονται στην Ιρλανδία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την καταστροφή του Συντηρητικού Κόμματο. Χαίρομαι που ο κύριο Τούς και ο κύριος Γιούνκερ δεν είναι εδώ, γιατί δεν ήταν καθόλου ήρεμοι και συχνά βάζουν τι προσωπικέ του προκαταλήψει πριν από τη διπλωματία. Πρέπει να το θυμάστε αυτό σε κάθε φορά που παίρνετε το λόγο. One minute, Mr. Μόνο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς, στις 21 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να συζητήσει μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό βλέπουμε όμως είναι ότι ε, ήδη από τον Ιούνιο θα υπάρχει ένας δασμός 25% όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε εδώ πέρα ότι η Γερμανία εφαρμόζοντας ένα μηδενικό συντελεστή δασμών ουσιαστικά θα υποφεληθεί περισσότερο από τις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα στραφεί κυρίως κατά των εξαγωγών της Γαλλίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κοινά πρότυπα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως θα επιβάλλουν και πάλι τα δικά τους τα πρότυπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να μειώσουμε όμως και τους γεωργικούς δασμούς. Αυτό απαιτούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει τελικά τι εκκλήσει τη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τελικά αν θα επικρατήσουν οι μεγάλε αυτοκινητοβιομηχανίε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αν αποφάσει αυτέ τελικά θα ληφθούν ει βάρο των Ευρωπαίων πολιτών που θα συνειδητοποιήσουν ότι οι αποφάσει αυτέ ισχύουν πάρα πολύ αργά. Ο κύριο Βαλίνσκι, για ένα λεπτό. Wer gestern im britischen Unterhaus die Debatte mitverfolgen konnte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 Κυρίες και κύριοι, όποιος παρακολούθησε χθε στη Βρετανική Βουλή Γινοτήτων τη συζήτηση ε, διαπίστωσε πόσο ε, μεγάλη διχόνοια υπάρχει στην Βρετανική πολιτική τάξη. Διχόνοια διότι υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία του Βρετανικού λαού που έδωσε μια σαφή εντολή. Μια εντολή αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει καμία σημασία αν ε, θεωρείτε ότι είναι καλή ή κακή αυτή η εντολή. Εάν εγώ θεωρώ ότι είναι καλή ή κακή. Είναι ένα θέμα σεβασμού. Σεβασμού της δημοκρατίας και των αποφάσεων που λαμβάνει η πλειοψηφία ενός λαού που έδωσε μια σαφή κατεύθυνση στην πολιτική της τάξη. Κάνω έκκληση. Σταματήστε αυτά τα τεχνάσματα. Σταματήστε από την πίσω πόρτα και από το παραθυράκι να οδηγήσετε σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Πρέπει να σεβόμεθα τις αποφάσεις ενός δημοψηφίσματος. Και θα την είχαμε σεβαστεί και αν είχαν ψηφίσει για την παραμονή. Τι θα γίνει, θα αλλάξει η στάση του Βρετανικού λαού και χρειαζόμαστε δεύτερο, δεύτερο δημοψήφισμα. Όχι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Εάν θέλουμε να παίρνουμε τον εαυτό μα σοβαρά και να μεταρρυθμίσουμε σωστά την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σεβόμαστε του κανόνε του παιχνιδιού και να δρούμε με υπεύθυνο τρόπο. Ευχαριστώ κύριο Συναρνός για ένα λεπτό. Βασιλείου δεν αποτελεί απλά ένα διαδικαστικό γεγονό. Σημαίνει ουσιαστικά την απόρριψη τη όποια σχεδιαζόμενη ομοσπονδοποίηση και την απαρχή μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αποτυπωθεί και στι επερχόμενε εκλογέ, Μια μετεξέλιξη βασιζόμενη στην άνοδο των υγιών πατριωτικών δυνάμεων με στόχο την ορθή λειτουργία τη Ένωση, όπω θα έπρεπε να υφίσταται επαναπατρίζοντα αρμοδιότητε υπό την κυριαρχία των κρατών μελών. Ο εκφοβισμό των εναπομεινάντων μελών δια του δίθεν παραγματικού τρόπου αντιμετώπισης του ηνωμένου βασιλείου θα καταρρεύσει. οι κρατούντες στην εξουσία τώρα αρνούμενοι να αποδεχθούν την εθελοντική και αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων κυρίαρχων κρατών αργά ή γρήγορα θα εξαναγκαστούν είτε σε απομάκρυνση είτε στο σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της έννοιας του κράτους έθνους. είναι καιρός να αναλάβουν σοβαροί άνθρωποι που υπηρετούν τους πολίτες ως πραγματικοί εκπρόσωποι απότοκος ευρείας συσπήρωσης και συνεργασιών πατριωτικών δυνάμεων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα για μια ευρώπη προσαρμοσμένη στα κράτη έθνη και όχι υποταγμένη στα οικονομικά συμφέροντα και την εξυπηρέτηση ολίγων και εκλεκτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Συμβούλιο Κομισιόν, κύριε Μπαρνιέ, εξαιρετική άψογη δουλειά που κάνατε. Η συμφωνία που επετεύχθη το βράδυ της Δευτέρας με την ε, Πρωθυπουργό κυρία Μέη ήταν μια ευκαιρία. Στην πραγματικότητα ήταν η ευκαιρία, η μοναδική ευκαιρία για να διευκολυνθεί μια εφτακτή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με εγγυήσει ε, προκειμένου ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να μην μείνει παγιδευμένο σε μια μόνιμη ταλωνιακή Ένωση αλλά απορρίφθηκε από την Βουλή από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, αυτό δείχνει έλλειψη ευθύνη. Ε, έλλειψη ευθύνη εκ μέρου μια πλειοψηφία βουλευτών ε, που μπλοκάρουν μονίμω μια λύση. Είναι κρίμα. Και είναι παράξενο που αύριο το ίδιο κοινοβούλιο θα ψηφίσει μια παράταση της παραμονής του Βασιλείου. Αυτό που δεν θα αλλάξει όμως με αυτό είναι οι όροι αποχώρησης. Οπότε αργά ή γρήγορα το νομο Βασίλειο θα πρέπει να πάρει την απόφαση τελικά ναι ή όχι σε μια συμφωνία. Αυτή είναι η ερώτηση. Και σε, αυτή την, σε αυτό το περιβάλλον ασάφειας ε, θα γίνουν εκλογές, ε, διάφορες εκλογές ε, ε, και επιλογές. Το το ζήτημα καταρχήν του αν θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, ε, διότι αυτό θα έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Δεύτερον, ε, το, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου σημαίνει ότι θα επηρεαστούν στην καθημερινότητά τους εκατομμύρια άνθρωποι σε πολύ καθημερινά πράγματα, μικρά και καθημερινά το πώς κανείς αγοράζει πιο φτηνά και πιο πολλά προϊόντα, ε, η ε, κάρτα ασφάλισης, ε, το κόστος του roaming και τρίτη επιλογή πρέπει να γίνει, τρίτο θέμα είναι η ρήξη, το ρήγμα που θα προκύψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός του Βασιλείου. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο σημαντική από ποτέ για, κάποια, για κάθε χώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Το να μην δρούμε μαζί από κοινού ε, μας εκθέτει, σε σημαντικ, εκθέτει σε σημαντικούς κινδύνους. Έχω ένα, μια άσχημη είδηση, κάποιοι θα εξοργιστούν μαζί μου, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με το Catch the Eye, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Η κυρία για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ορισμένε φορές ε, κατά τη διάρκεια των συνόδων εδώ πέρα στο Στρασβούργο α, αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις απογοήτευσης και ψευδεστήσεων. Μια τέτοια εβδομάδα αυτή τη στιγμή διανύουμε και αυτή τη φορά. Ακούσαμε του προαλήσαντε, ακούσαμε το αποτέλεσμα στην ψηφοφορία στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και συμφωνώ με πάρα πολλού συναδέλφου μου ότι όντω είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφανθεί εκ νέου ο Βρετανικό λαό. Υπάρχει πλήρε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο λαό είναι αυτό ο οποίο θα πρέπει να αποφανθεί και να σπάσει το αδιέξοδο αυτό. 60 νέοι άνθρωποι είχαν έρθει πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπάθησαν να πείσουν το Κοινοβούλιο να θέσει την κλιματική πολιτική ως σημαντική πρωταρχική προτεραιότητα. Και αυτό όχι μόνο επειδή το επίπεδο φιλοδοξίας για το 2030 είναι πολύ χαμηλό, ξέρετε ότι έχετε και μια συμφωνία μέχρι το 2030 την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε. Αν θέλουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε όμως στις δεσμεύσεις προβλέπονται η Συμφωνία των Παρισίων, τότε μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχουμε μειώσει εκμηδενήσει εντελώς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Χρειαζόμαστε λοιπόν το συντομότερο δυνατό μια νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Συμφωνία των Παρισίων να γίνει νομοθέτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να δεσμευτούν όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην υπάρχει παράβαση από κανένα κράτο. Αυτό ζητάνε οι νέοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλουν οι νέοι τη Υπήρου μα και πραγματικά θα λέγονται το μόνο αισιόδοξο μήνυμα που είχαμε αυτή την εβδομάδα. κύριο Σούλικη, ένα λεπτό παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Χθε είδαμε ότι υπήρξε ένα πραγματικό χάο στη Βουλή των Κοινοτήτων και βλέπουμε ότι η συμφωνία αποχώρηση είναι πλέον νεκρή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε επαοριστών. Δεν γίνεται να επιστρέφουμε πάντα στο σημείο 0. Ο χρόνο έχει τελειώσει. Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει βέβαια να γίνει σεβαστή. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη βούληση του Βρετανικού λαού. Γιατί αν κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε η στάση μα είναι ιδιαίτερα λανθασμένη το να προχωρήσουμε σε δεύτερο δημοψήφισμα είναι εντελώ ε, παράλογο, δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Μπορούμε να προετοιμαστούμε και η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να έχουμε ένα σκληρό Brexit, ένα Brexit χωρί συμφωνία αποχώρηση. Αν προσεγγίσουμε λοιπόν την όλη κατάσταση με νυφαλιότητα, τότε θα αρχίσουν να ισχύουν αυτόματα οι κανόνε του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Όταν και αν οι Βρετανοί πολίτε ζητήσουν παράταση αύριο, τότε εμεί μπορούμε να χορηγήσουμε την παράταση αυτή χωρί να υπάρχουν σημαντικέ δυσκολίε. Και σε αυτό το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τη παράταση μπορούμε να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικά βήματα προκειμένου να πετύχουμε τελικά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση η κλιματική αλλαγή θα, εξακολου... θα, θα είναι ξανά θέμα του, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα οξύμορο δίλημα. Κατα... Αφενός μειώνουμε τις εκπομπές, ε, Απ' την άλλη μεριά ενθαρρύνουμε ε, τι ε, ξέφρονε ελεύθερε συναλλαγέ κάτι που οδηγεί μηχανικά αυτόματα στην αύξηση των ίδιων αυτών εκπομπών. Οι συνθήκες ελεύθερων συναλλαγών μαζί με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν στην καταστροφή τη βιομηχανία μα. Και τι γίνεται, εισάγουμε ε, βιομηχανικά προϊόντα από άλλε χώρε που δεν έχουν τι ίδιε περιβαλλοντικέ, κοινωνικέ ε, και άλλε προδια... και υγειονομικέ προδιαγραφέ. Και όλα αυτά μετακινούνται με εμπορικά πλοία τεράστια τα οποία μολύνουν πολύ περισσότερο τη θάλασσα. Διοξίδιο, του θείου, οξίδιο του, διοξίδιο του άνθρακα κλπ. Μικροοργανισμοί, μικροσωματίδια κλπ. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το οικονομικό μα μοντέλο προστασία, επανεγκατάσταση και μικρέ αποστάσει να, να παράγουμε, να καταναλώνουμε και να ανακυκλώνουμε σε περιορισμένη γεωγραφική ακτίνα. Μόνο έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε τι οικολογικέ μα ανησυχίε με την οικονομία. Ευχαριστώ. Κύριε Χούμπνερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Η απόρριψη της συμφωνίας αποχώρησης ε, σημαίνει διάφορα πράγματα σημαντικά. Πρώτον, η έφτακτη αποχώρηση δύο εβδομάδες δεν θα γίνει. Δεύτερον, η προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν, καθώ επίση και η αποφυγή του συνόρου μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρεια Ιρλανδίας δεν επιτεύχθησαν και δεν πρόκειται να επιτευχθούν μέχρι το τέλο Μαρτίου. Η κίνδυνη είναι τεραστή Και αυτό είναι πολύ κακό. Αυτό είναι το, ε, τι θα γίνει αύριο με την ε, ψηφοφορία για την παράταση. Αν ψηφιστεί υπέρ της, ε, αν ψηφίσουν υπέρ της ε, παράτασης, πόσοι θα είναι αυτή η παράταση και για ποιο λόγο. Ε, μια μακρόχρονη παράταση θα δημιουργούσε πολιτικά και εκλογικά προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσει και προβλήματα διαπραγμάτευσης στο μέλλον. σε κάθε περίπτωση η συμφωνία δεν θα ξανανοίξει. Με μακρά παράταση σημαίνει μακρότερη περίοδο αβεβαιότητας. Το νούμερο έχει πει πόσο σημαντικό είναι, η σημαντική είναι η έφρακτη αποχώρηση εδώ και πολύ καιρό και επανειλημμένος. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί άλλωστε εμπιστοσύνη στι διαπραγματεύσει για μια μελλοντική δίκαιη σχέση. Και αυτό θα πρέπει να το επαναλάβουμε και σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φαγιόν, ένα μισή λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφε, οι αρχοί κρατών και κυβερνήσεων ε, θα συζητήσουν για την οικονομία αλλά πρέπει να συνδέασουμε την ε, οικονομία με το περιβάλλον και να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας. Αυτό μας λένε οι νέοι και οι λαοί. Μετά την ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο μπορούμε μόνο να ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει σκληρό Brexit. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε την τελευταία συνάντηση κορυφής πριν από τις ευρωεκλογέ. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ευθύνη. Οι πολίτες αναμένουν δράση, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα δράξουμε και πάλι την ευκαιρία. Ας σκεφτούμε πόσο έχει αποτύχει η διαχείριση τη μετανάστευση. Εμείς εγκρίναμε όλους τους κανόνες που είναι αναγκαίοι για να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευση και ασφαλέστερα σύνορα. Αλλά τα κράτη-μέλη και διάφοροι εθνικιστέ πολιτικές έχουν την ευθύνη. Σε αυτού πρέπει να, ε, πρέπει να καταδείξουμε σαφώ ω υπευθύνου. Διότι είναι γνωστοί οι λόγοι που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα είναι ο λαϊκισμός. Ε, ο καθένας προσπαθεί με λαϊκιστικά επιχειρήματα να ρίξει την ευθύνη στους άλλους. Αγνοούν οι ηγέτες μας την ε, ανησυχία των λαών. Εδώ και πέντε χρόνια μας λένε οι πολίτες μας ότι είναι η μεγαλύτερη ανησυχία τους. Πώς θα πάμε τώρα στις ε, κάλπες. Το βασικό είναι να υπάρξει μια κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη που να αντιμετωπίζει τα ψεύδι τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό. Πρέπει πραγματικά να επιδιώξουμε να υπάρχει ένα άλλο μέλλον για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ κυρία Τόμασιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το Brexit ε, έχει γίνει ένα πραγματικό χάος. Αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε από την ε, πλευρά των Βρυξελών καλή πίστη. Εμείς ε, στις Βρυξέλλες δηλαδή επιδιώξαμε να αποδείξουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα και ευημερία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Βρετανοί προσπάθησαν να επιτύχουν το αδύνατο να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή σε αυτήν. Η περίπλοκη πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο έκανε ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση και έγινε ακόμη πιο περίπλοκη από τις δύο πλευρές και δεν είναι δυνατόν τελικά να υπάρξει μία ε, συντεταγμένη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι διαπιστώνουμε, ο καθένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, ενώ ευθύνε έχουν και οι δύο πλευρέ. Δεν πρέπει να επανέλθουμε στο παρελθόν, πρέπει να στραφούμε προ το μέλλον. Θα πρέπει να μπορούμε να συνεργαστούμε στα βασικά σημεία και να έχουμε εμπορικέ συναλλαγέ χωρί ε, προσκόμματα, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Νίτερμαερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση για τον Brexit. Η λεγόμενη κακή συμφωνία δεν ε, ήταν αντικείμενο της διαπραγμάτευσης ε, από την πλευρά του κ. Μπαρνιέ αλλά και από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόβλημα δεν είναι η συμφωνία, είναι η πολιτική κρίση που διαπιστώνουμε στο Λονδίνο και η οποία υποδαβλίστηκε από πολλούς που πήραν το λόγο εδώ σήμερα και μετά σκόθηκαν και έφυγαν, ως συνήθως. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα. Γι' αυτά θέλω να μιλήσω. Με τα οποία πρέπει να αποσχοληθεί η συνάντηση κορυφή. Τα οικονομικά θέματα. Μετά του ε, καλού καιρού μπορεί να έχουμε λιγότερο καλού καιρού που μπορεί να πυροδοτηθούν από του εμπορικού πολέμου, τον Brexit ή άλλα γεγονότα. Άρα τα κράτη-μέλη πρέπει να δουν πόσο ρωμαλαίες είναι οι οικονομίες μας, πόσο προετοιμασμένες είναι για επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και ίσως και άλλα ε, αρνητικά γεγονότα. Το δεύτερο σημαντικό για μένα είναι η Κίνα. Πιστεύω ότι έναντι της Κίνας πρέπει να είμαστε πιο κατηγορηματικοί, πρέπει να τονίσουμε πιο πολύ ότι έχουμε ε, νόμιμα συμφέροντα και να είμαστε πιο ε, στεναρείς διαπραγματεύσεις. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ο κινέζικος νόμος για την ε, κυβερνοασφάλεια. Και έχουμε και άλλα μεγάλα θέματα. Όπω ε, η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να συμμετάσχει και η Κίνα στην επίλυση του θέματο αυτού και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Βάιντενχολτσα. Ένα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Μα είναι τραγικά αυτά. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα κράτο που είναι δικαίω περήφανο για την ιστορία του, και που έχει ε, βοηθήσει αλλά και βοηθηθεί πολύ από την Ευρώπη αυτοδιαλύεται και γίνεται και γελίο. Δεν έχουν κατεύθυνση, δεν έχουν ε, πολιτική βούληση, κινδυνεύουν πραγματικά να καταρρεύσουν. Και αυτά τα παρατηρούμε ε, με αμηχανία αλλά και εκνευρισμό. Μία ολόκληρη γενιά θα θυγεί από τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης. Σε αυτήν την ιστορική στιγμή δεν πρέπει να κάνουμε επιπλέον λάθη πρέπει να έχουμε μια στενή ε, σχέση με τους Βρετανούς που να βασίζεται σε αυτό που υποτίθεται πάσχουν και οι Βρετανοί, πραγματισμό. Πρέπει να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στους Βρετανούς φίλους. Οποιαδήποτε άλλη ε, ε, επιλογή θα ήταν υπεροψία. Νομίζω ότι η παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι, όπως και πριν, η καλύτερη λύση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει νομιμοποιούμενο με ένα δημοψήφισμα, το οποίο αντίθετα με το προηγούμενο πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να υπάρξει σαφήνεια για τα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών στην, ε, στο Ενωμένο Βασίλειο και τα 1,3 ε, που είναι ε, στο των Βρετανών πολιτών που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ε, μεγάλη αγωνία. Τα άτομα αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν παιχνιδάκι στην πολιτική διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό. Οι δραματικές εξελίξεις με αφορμή το Brexit κλειδονίζουν τη γυραιά Ήπειρο. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το Brexit έστειλε ένα μήνυμα ισχυρό. Ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί αναζητούν ένα άλλο δρόμο για την Ευρώπη μια ευρώπη των εθνών και των πατρίδων μια ευρώπη που να σέβεται τις εθνικές παραδόσεις και τους λαούς μια ευρώπη δημοκρατική και αποκεντρωμένη μια ευρώπη της αλληλεγγύης και όχι του σκληρού πυρήνα μια κοινωνική ευρώπη και όχι μια ευρώπη των τραπεζών. οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν αντέχουν τη λιτότητα και τη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που έχουν επιβάλει το eurogroup και η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και σύντομα θα στείλουν ισχυρό μήνυμα στις επικείμενες ευρωεκλογές γιατί για την ευρώπη υπάρχει άλλος δρόμος ο δρόμος της ανάκτησης της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών της ο δρόμος ενάντια στην κινεζοποίηση των μισθών ο δρόμος ενάντια στη γερμανική ευρώπη. Κυρία Γκέρλινγκ, λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χθε το βράδυ είδαμε μία ακόμη φορά ότι το Βρετανικό Κοινοβούλιο δεν καταφέρει να καταλήξει σε συνένεση. Μια μειωμένη πλειοψηφία που όμως παρόλα αυτά οδήγησε σε δεύτερη συντριπτική πλειοψηφία σε ψηφοφορία στην ιστορία του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Τρεις είναι οι επιλογές που έθεσε χθε η κυρία Μέη. Ανάκληση του άρθρου 50 καταρχάς. Πρώτη φορά προφέρει δημοσίως κάτι τέτοιο. Δεύτερον, αναφέρθηκε στην διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι ε, ανέφερε ίδια τις λέξεις αυτές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τρίτον, πραγμάτευση ενός μιας νέας συμφωνίας. Νομίζω ότι η τρίτη επιλογή δεν είναι σε λογικά χρονικά περιθώρια τουλάχιστον εφικτή. Άρα αυτή τη στιγμή που έχουμε δύο επιλογές, no deal ή no Brexit. Νομίζω ότι το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα καταψηφίσει το no deal, αλλά όχι το no Brexit. Έχουμε περιορισμένο ρόλο εδώ πέρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη διατύπωση των παρεμβάσεών μα. Στέλνουμε κάποια μηνύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια ισχυρή βούληση στον Ηνωμένο Βασίλειο για δεύτερη ψηφοφορία. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί θέλουν δεύτερο δημοψήφισμα και οι δημοσκοπήσει δείχνουν ότι πολλοί θέλουν το δεύτερο αυτό δημοψήφισμα. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο να διοργανωθεί κάτι τέτοιο, αλλά μην ακούτε μην πιστεύετε αυτά τα οποία είπαν σήμερα Βρετανοί συνάδελφοι. 7, από τους 9 βουλευτές στην αίθουσα αυτή ουσιαστικά αντιστοιχούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Δεν είναι αυτοί οι πατριώτες, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν ένα no deal Brexit. Α μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή τα όσα λένε στρέφονται κατά του Βρετανικού λαού και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πατριώτε, κανεί δεν του αποκαλεί έτσι. Κανεί δεν θα ήθελε ουσιαστικά να προωθηθεί η δικιά του συστάση, η οποία μπορεί να είναι τόσο επιζήμια. Κανεί ο οποίο θέλει να υποστηρίξει τη συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή, ποτέ δεν θα ήθελε ένα Brexit χωρί συμφωνία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στην πλειοψηφία βρίσκονται στο περιθώριο θα έλεγα, πηγαίνουν στο μπαρ του κοινοβουλίου, δεν συμμετέχουν καν στις δημόσιες συνεδριάσεις, δεν ακούνε αυτά τα οποία λένε οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Επομένως είστε παροχημένε πλέον φωνέ είστε φωνέ φωνές του χθε. Εμείς και άλλοι συναδελφοί μου, ομοειδάτε με μένα, εκπροσωπούν τη φωνή του σήμερα και του αύριο. Σκόρμπετ για δύο λεπτά. Μετά την πρώτη απόρριψη της ε, συμφωνίας τον Ιανουάριο, η Τερέζα Μέη προσπάθησε να επαναδιαπραγματευτεί ένα μόνο σημείο, το backstop της, ε, για την Ιρλανδία προκειμένου να εξευμενήσει τη δεξιά πτέρυγα του, του κόμματό τη. Όμω για την πλειοψηφία στην ε, Βουλή των Κοινοτήτων δεν ήταν αυτό το βασικό πρόβλημα. Υπήρχαν άλλα προβλήματα τα οποία η κυρία Μέη δεν προσπάθησε να αντιμετωπίσει προσπάθησε να επιλύσει, ε, να εξευμενήσει μόνο την ε, δεξιά πτέρυγα του κομματό τη. Οπότε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πλειοψηφία στην πολιτοκοινοτήτων δεν θέλει να βγει η, Βρετανία χωρί συμφωνία. Αλλά η μόνη συμφωνία που υπήρχε έχει απορριφθει Οπότε πού βρισκόμαστε. Δύο δυνατότητε προφανώ. Ή διαπραγματευόμαστε μια δεύτερη συμφωνία ή ξαναθέτουμε σε συζήτηση το Brexit. Ε, αυτό όμως, ε, ε, η πρώτη λύση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η δεύτερη λύση απαιτεί δεύτερο δημοψήφισμα. Και όπως είπε η κυρία Γκέρλινγκ, υπάρχει μια πλειοψηφία στην κοινή γνώμη που επιζητεί, επιθυμεί ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Και οι δημοσκοπήσεις λένε ότι αν γίνει δεύτερο δημοψήφισμα, ο λαός θα ψήφιζε παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε θα ήταν τρέλα να συνεχίσουμε με τον Brexit, λέγοντας χειριζόμενοι ότι αποτελεί βούληση του ε, του λαού. Αξίζει να δούμε αν ο λαός πράγματι επιμένει σε αυτό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρας, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σαφές για όλους μας. Ε, αν δεν αλλάξει η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 29 Μαρτίου, θα υπάρξει χαοτική, σκληρή αποχώρηση. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι όποιος δεν θέλει να απευθυνθεί διακομματικά δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, τα οικονομικά, τα οικολογικά, τα κοινωνικά, τα τεχνολογικά, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις προκλήσεις για δημοκρατία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από κοινού στην Ευρώπη. Διακομματικά με την συνεργασία όλων των ε, δυνάμεων για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της Ευρώπης στον κόσμο. Περί αυτού πρόκειται στι ευρωεκλογέ και περί αυτού πρόκειται για τη σύσταση τη επόμενη επιτροπή. Και αυτή η πραγματικότητα είναι σε απόλυτη αντίφαση με την πολιτική αποτυχία των πολιτικών υπευθύνων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά και σε άλλα πολιτικά κόμματα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε τι γίνεται στην Σλοβακία, όπου, και τη Μάλτα όπου δολοφονούνται δημοσιογράφοι, την κατάσταση με το κράτος δικαίου στην ε, Ουγγαρία και την Πολωνία, την αύξηση στην Ουγγαρία, την Ιταλία, την Τσεχία και την Ρουμανία των ε, λαϊκιστικών και εθνικιστικών δυνάμεων. Τα ευρωπαϊκά ιδεώδη υπονομεύονται εκ των έσω. Αυτή η εκ των έσω υπονόμευση πρέπει να αντιμετωπιστεί στις ευρωεκλογές με το να ψε, λέμε ψέματα, τον, τον αντισημιτισμό, τον εθνικισμό και με το να κατηγορούμε ένα τον άλλον και την απομόνωση δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα στην Ευρώπη, ούτε το Brexit. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα μορφή βασικής συνένεσης. Ο κύριος Κέλλη, 1,5 λεπτό. Μετά την απόρριψη της συμφωνίας απόρριψης από την Βουλή των Κοινοτήτων χθες το βράδυ, υπάρχει πολύ φόβος στην Ιρλανδία, ανησυχία ιδιαίτερα μεταξύ των γεωργών και του αγροτροφημικού τομέα. Ξέρουν ότι μία σκληρή αποχώρηση σύνορα και η χρήση των κανόνων του ΠΟΕ θα τους χρεοκοπήσουν. Ξέρουμε ότι αν υπάρξει σκληρή έξοδος, η ειρήνη που έχουμε τα τελευταία χρόνια και που κατακτήσαμε με τόσους αγώνες θα κινδυνεύσει. Γι' αυτό ελπίζω σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων να υπερψηφιστεί η απόρριψη ενός σκληρού Brexit, μιας άτακτης αποχώρησης. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει αυτομάτως να τους προσφέρουμε μια παράταση, χωρίς προϋποθέσεις. Πρέπει να τους την προσφέρουμε. Μπορούμε να το κάνουμε για τρεις μήνες, χωρίς ε, να ε, επηράσουμε κατά κανένα τρόπο τις εκλογές. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ας τους βοηθήσουμε να βρούνε κάποιο άλλο τρόπο. Και ίσως αυτός ο άλλος τρόπος να είναι η παραμονή. Δεν θα ήταν αυτό. Δεν θα ήταν αυτό κάτι που πραγματικά πρέπει να το επιθυμούμε. Και δεν θα βοηθούσε μια παράταση σε κάτι τέτοιο. Κάνω έκκληση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει καλόπιστα. Να πει ναι, ναι θα σας βοηθήσουμε. Θα σας δώσουμε το χρόνο που χρειάζεστε. Ούτως ώστε να τακτοποιήσετε τα του οίκου σας να αποφύγουμε ένα σκληρό Brexit, να αποφύγουμε μια άτακτη αποχώρηση. Εάν σοβαρά θέλετε να βρείτε μια άλλη λύση, θα σας το επιτρέψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σουίτσα τώρα για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι ε, η συζήτηση για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει γίνει περισσότερο συζήτηση για τον Brexit αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε όπω θα έπρεπε για τι πράσινε τεχνολογίε για τη Συμφωνία των Παρισίων. Δεν συζητάμε για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ούτε καν για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την παραπληροφόρηση που μα βάλει από όλε τι πλευρέ. Δυστυχώ, η συζήτηση που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή είναι μια συζήτηση για τον Brexit. Προφανώ το Brexit είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή σε αυτά τα οποία θα πρέπει να συζητάμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης. Ακούσαμε όλους αυτούς που αναφέρθηκαν σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για ένα δεύτερο δημοψήφισμα στον Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό διότι πιστεύω ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ειλικρινά λυπάμαι που οι λαϊκιστές ε, έχουν νικήσει τελικά στο δημοψήφισμα, στο προηγούμενο δημοψήφισμα. Πιστεύω όμως ότι αυτό μπορεί να τροποποιηθεί. Πιστεύω ότι ε, οι Βρετανοί πολιτικοί θα αναλάβουν τις ευθύνε του και θα συνειδητοποιήσουν πω έχει πραγματικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή και δεν θα υπονομεύσουν σε καμία περίπτωση το μέλλον των νέων, των νέων εκείνων οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. έχει το λόγο, δεδομένου ότι οι υπομιλητές ε, ολοκλήρωσαν τις παρεμβάσεις τους. Κ. σε ευχαριστώ πολύ. Άκουσα πολύ προσεκτικά το Κοινοβούλιο. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πολύ ευρεία στήριξη ε, του τρόπου με τον οποίο η Κομισιόν διεξάγει διαπραγματεύσει ε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών Μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσπαθώντα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για μια συμφωνία αποχώρηση που θα βλάψει όσο το δυνατό λιγότερο και τι δύο πλευρέ. Αυτή ήταν άλλωστε και η πρόθεση τη Κομισιόν εξ αρχή. Αυτό ήταν ο τρόπο με τον οποίο ο Μισελ Μπαχνιέ διεξήγαγε τι διαπραγματεύσει από την αρχή. Και ενισχύεται η θέση μας μετά την σημερινή συζήτηση. Έχοντας ακούσει τον κύριο Φαράτζ και τους ε, συναδέλφους του και έχοντας ε, διαπιστώσει την τεράστια ύβρη με την οποία φέρεται, με την και αυτή στάση την οποία επιδεικνύει, αναρωτιέμαι μερικές φορές. Έχει πάει στο Σάντερλαντ να μιλήσει με τους εργάτες του εργοστασίου της Νισάν και να τους πει θα μπορεί να σας κοστίσει την ε, δουλειά σας, αλλά εγώ θα κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου. Πήγε, πήγε στην Οξφόρδη.